Ladies Κυρίες και κύριοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε την συνεδρίαση σήμερα το απόγευμα. Είναι 3, και 36, έχουμε αργήσει λίγο. Έχω να σας ενημερώσω για τα εξής. Η κυρία Νικόλη Σόνοβα δυστυχώς δεν μπορεί να προεδρεύσει σήμερα και ακριβώς επειδή η μερίσια διάταξη είναι πάρα πολύ μεγάλη και δύσκολη θα ήθελα να μιλήσω τη γλώσσα μου, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Ωραία λοιπόν, ξεκινάει η συνεδρίαση. Πάμε στο πρώτο σημείο. Μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μέχρι το τέλος συνεδρίασης. Έχει κάποιος ε, κάποια αντίρρηση, ένσταση. Μάλιστα. Μετά. Διερμηνία υπάρχει σε πάρα πολλές γλώσσες, σχεδόν σε όλες, εκτός από τα μαλτέζικα. Σημείο 3. Πρακτικά. Εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις που δεν βλέπω να υπάρχουν, μπορούμε να εγκρίνουμε τα πρακτικά. Και τώρα περνάμε στο σημείο 4 και τους προσκεκλημένους μας σήμερα. Καλωσορίζω λοιπόν τον κύριο Χάιντς Μπέκερ, ο οποίος είναι υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΤΕΦΟΠ. Στη συνέχεια καλωσορίζω την κυρία Βερόνικα Λόπε Φοντανιέ. από την Eurofound. Και οι δύο επόμενοι καλεσμένοι μας σήμερα, στα δεξιά μου, είναι ο κύριος Μίξιτς για την EU OSHA και ο κύριος Γιάν Κρέμερς για την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας. Βρίσκεστε όλοι εδώ, χαίρομαι πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Έχω να προτείνω το εξής. Εάν δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση, μπορούμε να ακούσουμε τους προσκεκλημένους μας στη σειρά και μετά να ξεκινήσει ο γύρος των ερωτήσεων. Κατά τον πρώτο γύρο ερωτήσεων, όπως γνωρίζετε, θα λάβουν το λόγο οι συντονιστές και συντονίστριες, ο καθένας από δύο λεπτά, έτσι ώστε να θέσουν τις ερωτήσεις τους στους υποψήφιους. Και κατόπιν θα περάσουμε στο δεύτερο κύκλο ερωτήσεων, δεύτερο γύρο όπου θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν το λόγο οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές εφόσον το επιθυμούν. Έπειτα, όπως βλέπετε, το σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης, που θα εξεταστεί στις 5 περίπου, αφορά τις ψηφοφορίες. Όμως, μπορούμε να ξεκινήσουμε με τις παρουσιάσεις των υποψηφίων. Και πρώτος θα λάβει το λόγο ο κύριος Μπέκερ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα κάνω την παρουσίασή μου στα γερμανικά, διότι δεν θα ήθελα να υποστείτε την αυστριακή μου προφορά. Είναι μεγάλη μου τιμή, λοιπόν, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να παρουσιάζομαι σήμερα ενώπιόν σας ως υποψήφιος ε, εμπειρογνώμονας για την ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτήν την τιμή. Πολλοί από εσά ίσω γνωρίζετε ότι υπήρξα ευρωβουλευτή μέχρι τον Ιούλιο φέτο του 2019. Και από το 2011 ήμουν μέλος της Επιτροπής σας. Τακτικό μέλος και αναπληρωματικό μέλος, καθώς και αναπληρωτής συντονιστής. Με την ιδιότητα αυτή υπήρξα πολύ ενεργός. Επίσης υπήρξα εισηγητή σε πολλούς ε, σημαντικούς φακέλους καθώς και σκιώδης εισηγητής ε, για θέματα τα οποία μας αφορούν. Για παράδειγμα την έκθεση για το Γιούρες, την πρωτοβουλία για την κοινωνική οικονομία και την οικονομία αλληλεγγύη, στη Λευκή Βίβλο για τις συντάξεις και πρόσφατα την ε, ανακατάταξη των ευρωπαϊκών υπηρεσιών. Ήμουν λοιπόν εισηγητής ή συνεισηγητής αυτές τις εκθέσεις. Από το 2005 είμαι μέλος του Προεδρείου ε, του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην Αυστρία και στην παρουσίασή μου σήμερα θα ήθελα να σας ε, αναφέρω τις ιδέες μου και τις ελπίδες μου για την υποψηφιότητά μου. Έχω καλή γνώση πάνω στα θέματα επαγγελματικής κατάρτισης ε, και λόγω της ιδιότητάς μου ως ε, μέλος της, Ευρωπαϊ... Επιτροπής Απασχόλησης ε, είχα δώσει βάση στην καταπολέμηση της ανεργίας, ειδικά της ανεργίας των νέων και υπήρξα μέλος αρκετών πρωτοβουλειών. Πάντα με ενδιέφερε το ζήτημα των επαγγελματικών προσόντων. Μετά ασχολήθηκα με την εγγύηση για τους νέους, με διάφορα θέματα σχετικά με την αγορά εργασίας. Και απέκτησα λοιπόν σημαντική εμπειρία. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ευρωπαϊκός ε, πυλώνας των κοινωνικών δικαιωμάτων. Είναι ένα κατόρθωμα που προέκυψε μετά από κόπους αιώνων και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εξακολουθεί να είναι σημαντικό ακόμα και σήμερα. Έχουμε δει ότι έχουμε καταφέρει πολλά, πολλά περισσότερα από όσα ονειρευόμασταν. Όμως σίγουρα μας μένουν πολλά ακόμα να πραγματοποιήσουμε. Ως μέρος της υποψηφιότητάς μου θεωρώ πως ε, μπορώ να εκπροσωπήσω τα συμφέροντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Απασχόλησης. Η εμπειρία που αποκόμισα με κάνει να πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα η Επιτροπή Απασχόλησης εκτιμούν ιδιαίτερα τον ρόλο που διαδραματίζουν οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες και οι ευρωπαϊκοί αυτοί οργανισμοί. Αυτό είναι που μου έδωσε και το κίνητρο να θέσω υποψηφιότητα για μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Και παρότι ο ρόλος του εμπειρογνώμονα δεν ε, έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Θα ήθελα να ασχοληθώ με θέματα τα οποία με εκφράζουν ιδιαίτερα και με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Τόσο η ΣΕΝΤΕΦΟ όσο και οι άλλες ευρωπαϊκές υπηρεσίες οι οποίες ε, συνεργάζονται και ασχολούνται με παρόμοια θέματα νομίζω πως ε, έχουν μεγάλο δυναμικό και εμείς οφείλουμε να ασκήσουμε πίεση μέσω των υπηρεσιών αυτών, μέσω των, της ιδιότητάς μας, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τις, ε, να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και να εφαρμόσουν τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οδηγίες. Οπωσδήποτε πρέπει να ασκήσουμε την ήπια δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς. θεωρώ ότι τα διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα ή διαφορετική κουλτούρα σε ό,τι αφορά την επαγγελματική ε, κατάρτιση στα κράτη-μέλη χρειάζεται έναν συγχρονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε να υπάρξει μία προσέγγιση των διαφορετικών ε, στοιχείων τους. Δεν σημαίνει αυτό απαραίτητα ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο, όμως η εκπαίδευση δύο κατευθύνσεων, όπως ε, λειτουργεί αυτή τη στιγμή στη Γερμανία και την Αυστρία, είναι μια καλή ιδέα. Δεν σημαίνει βέβαια ότι, θα, ότι πρέπει να εφαρμόσουμε κατά γράμμα το αυστριακό και γερμανικό πρότυπο, όμως πιστεύω ότι μπορούμε να αντλήσουμε ιδέες. Χρειάζεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές για να τεθούν κάποια κεντρικά σημεία στα οποία πρέπει να δώσουμε βάρος. Η Ευρώπη των 27 αλλά και οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι φορείς έχουν λοιπόν μεγάλο έργο μπροστά τους. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει ένα σαφής ορισμός της απασχολησιμότητας, employability στα αγγλικά, και να δοθεί έμφαση ιδιαίτερα στην απασχολησιμότητα των νέων αλλά και των ε, ηλικιωμένων, οι οποίοι έχουν ψηλά ποσοστά ανεργίας. Αυτή λοιπόν η απασχολησιμότητα νομίζω πως θα πρέπει να είναι πάντα το κύριο μέλημά μας. Πρέπει να δούμε αν μπορούμε να τηρήσουμε τις ε, δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό, νομίζω πως θα πρέπει να δοθεί έμφαση στις ψηφιακές τεχνολογίες. Αυτό είναι προφανές. Έχουμε παρατηρήσει ότι υπάρχει αυξημένη κινητικότητα στην αγορά εργασίας, αλλά θεωρώ πως χρειάζεται βελτίωση στην κατάρτιση δασκάλων και εκπαιδευτών. Ακριβώς διότι από τις πληροφορίες που έχουμε δεν ε, πληρεί τις ε, προϋποθέσεις ποιότητας που έχουν τεθεί. Επίσης, οι νέοι είναι πολύ σημαντικοί. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα ε, της ε, εκπαίδευσης και κατάρτισης των νέων. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε τους νέους έτσι ώστε να μην εγκαταλείπουν το σχολείο, έτσι ώστε να έχουν τα εφόδια για να βγουν έπειτα στην αγορά εργασίας. Όχι όμως ε, μόνο οι νέοι, αλλά όλες οι ηλικιακέ ομάδες και οι ηλικιωμένοι. Θεωρώ ότι ένας συνδυασμός νέων και μεγαλύτερων ενηλίκων σε ομάδες νομίζω πως θα βελτιώσει την κατάσταση. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό για μένα να μειωθεί η, διαφο η μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών. Έχουμε εξάλλου ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίσει και την αντίστοιχη έκθεση. Επίσης, πολύ σημαντική είναι και η ένταξη των ε, μεταναστών και των ε, τον άσυλο στην αγορά εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ επίσης ότι η κοινωνική οικονομία της ε, Ευρώπης, ένα θέμα το, για το οποίο ήμουν και εισηγητής, θα είναι η κινητήριος δύναμη σε ό,τι φορά τα θέματα επαγγελματικής κατάρτισης. Θα ήθελα να κλείσω την παρουσίασή μου με το εξής. Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΝΤΕΦΟΠ έχει δώσει ένα σύνθημα στις 24 Σεπτεμβρίου. Πρέπει δηλαδή να εξοπλιστούμε και να είμαστε έτοιμοι για το μέλλον. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε και εδώ θα σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ και μπορούμε να συνεχίσουμε με την κυρία Βερόνικα Φοντανιέ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα μιλήσω σπανικά. Να πω ότι είναι κάπως ε, παράξενο για μένα μετά από δύο θητείες ε, ως ε, βουλευτής και μάλιστα στην Επιτροπή Απασχόλησης να βρίσκομαι εδώ και μπορώ να πω ότι είναι τιμή μου να βρίσκομαι εδώ ενώπιόν σα ω ε, υποψήφια εμπειρογνώμονα ε, για το EuroFound, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα τη Βελτίωση Συνθήκων Διαβίωση και εργασία. Είναι πολύ ιδιαίτερη αυτή η επιτροπή και η αλήθεια είναι ότι εγώ πιστεύω ότι πάντοτε έκανε πολύ καλή δουλειά και υπήρχε και μεγάλη σύμπνοια. Έχω πάρα πολύ καλέ αναμνήσεις. Τώρα, ποιος ε, θα είναι ο ρόλος του εμπειρογνώμονα στο Eurofound. Εγώ θα σας πω πώς το σκέφτομαι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει και μπορεί να κάνει περισσότερα για τους πολίτες. Κάθε πολίτης μετράει και πρέπει να έχουμε προσωποποιημένη εστίαση για όσους ε, βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης. Το Eurofound μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμο για να το πετύχουμε. Από τη δημιουργία του το 1975, Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Βελτίωση Συνθήκων Διαβίωσης και Εργασίας, έχει συνεισφέρει στην προώθηση της βελτίωσης ε, των συνθήκων ζωής και εργασίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσφέροντας ε, γνώσεις εμπειρικής βάσης που επέτρεψαν οι κοινωνικές και εργασιακές πολιτικές να βασίζονται σε αντικειμενικά δεδομένα. Με αυτόν τον τρόπο οι εθνικοί και ευρωπαίοι πολιτικοί θύνοντες όπως και οι κοινωνικοί εταίροι και οι διεθνείς οργανισμοί μπορούν να γνωρίζουν ε, με μεγαλύτερη ακρίβεια ένα πιθανό πρόβλημα έτσι ώστε να μπορούν να βρεθούν κοινέ οικονομικές ε, και κοινωνικές λύσεις που να είναι βιώσιμες. Πρέπει να αναγνωρίσω τη σημαντική δουλειά που γίνεται καθώς ε, και τη χρησιμότητα των στοιχείων αυτών για τους Ευρωπαίους νομοθέτες. Καθώς και εγώ ίδια, βάσει της δικής μου εμπειρίας, τους χρησιμοποίησα τα δεδομένα αυτά πολλάκις τα τελευταία έτη. Γι' αυτό σας συνιστώ να τα χρησιμοποιήσετε και στο δικό σας έργο γιατί είναι κάτι πολύ χρήσιμο. Επίσης, συνειδητοποιώ πλήρως ε, τη δουλειά που υλοποιεί η Επιτροπή αυτή και τις ε, ανησυχίες της. Για το λόγο αυτό, στην ε, περίπτωση που εγκρίνεται την υποψηφιότητά μου, δεσμεύομαι η φωνή της Επιτροπής Απασχόλησης να ακούγεται όπως ε, πρέπει, όπως είναι πρέπον μέσα στο Eurofound. Και θα υπάρχει μια πολύ σημαντική σχέση μεταξύ των δύο. Πέρα από την πρόοδο που έγινε προς μια οικονομική και κοινωνική σύγκληση μεταξύ των διάφορων ε, κρατών μελών τις τελευταίες δεκαετίες, η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση προκάλεσε ένα τέλμα και ακριβώς αυτές οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες εξακολουθούν να υπάρχουν σε κράτη-μέλη και αυτές δημιουργούν εμπόδια στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης που αποτελεί τη βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης και εργασίας των Ευρωπαίων πολιτών. Επομένως, θα πρέπει να εργαστούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορέσουμε να αυξήσουμε την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα. Ενώ ταυτόχρονα θα εγγυόμαστε μία βιώσιμη αύξηση της απασχόλησης μία αύξηση των επεπίδων απεσχόληση που δεν θα πρέπει να επικεντρώνεται ε, σε ποσοτικούς όρου αποκλειστικά, αλλά θα πρέπει να γίνεται και με ποιοτικού όρου, καθώ το μελλοντικό ευρωπαϊκό μοντέλο δεν μπορεί να βασίζεται σε χαμηλού μισθούς. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου πως ε, οι μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες προοπτικές οικονομικό επίπεδο δεν είναι πολύ ευίωνες και οι εμπορικές εντάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως μεταξύ ΙΠΑ και Κίνας, ε, η οικονομική επιβράδυνση που βλέπουμε στη Γερμανία και στην Ιταλία ε, τα προβλήματα του μεταπητικού τομέα ή το τι θα γίνει μετά το Brexit, οι άγνοι αυτοί, απειλούν την ανθεκτικότητα των εθνικών οικονομιών και επομένως ε, της κατάσταση της αγοράς. Επομένως είναι σημαντικό να είμαστε προετοιμασμένοι για μια πιθανή έλευση κρίσης και να ενισχύσουμε το μίσο όπως η κοινωνική οικονομία. Υπό την έννοια αυτή οι επιχειρήσεις και πρέπει να αναγνωρίσω γιατί εργαστήκαμε πολύ στην προηγούμενη θητεία στο θέμα αυτό. Εργαστήκαμε με τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας και είδαμε ότι πέρα από το ότι ε, ευρωούν ε, την ε, συμπερίληψη κάποιων ευάλωτων ομάδων και μας έδειξαν ότι δεν έχασαν θέσεις απασχόλησης, αλλά κατόρθωσαν και να δημιουργήσουν μάλιστα. Αυτό έγινε με τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας. Επίσης πρέπει να έχουμε κατά νου ότι εμφανίζονται νέες προκλήσεις ε, λόγω της αυξανόμενης ανησυχίας για το περιβάλλον. Την δημογραφική αλλαγή πέρα από την κυρίανση του πληθυσμού και ιδίως ε, η ψηφιακή εποχή και ε, η τεχνολογική επανάσταση θα έχουν συνέπειες στις εργασιακές σχέσεις όπως τις γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Για να μπορέσουμε με επιτυχία να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις, είναι σημαντικό οι νομοθέτες να έχουν τα κατάλληλα δεδομένα προκειμένου να μπορέσουν να εξορροπήσουν τα αιτήματα των επιχειρήσεων και των εργαζομένων και της κοινωνίας, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της να υποφεληθεί από τα πλεονεκτήματα της ψηφιοποίησης, ενώ θα ελεγχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι που προκύπτουν από αυτή. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι πολίτες μας είναι το μεγαλύτερο ενεργητικό που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένως θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των πολιτικών μας. Μόνο με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να πετύχουμε μια κοινωνία ισότιμη οι νέες μορφές απασχόλησης ε, που δημιουργούνται λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης ε, ε, ζητούν περισσότερη ευελιξία και προσαρμογή των εργασιακών σχέσεων. Γι' αυτό όμως το λόγο δεν πρέπει να εξελιχθούν δικαιώματα. Οι εργάτες στις πλατφόρμες πρέπει να έχουν την κατάλληλη ρύθμιση και θα να υπάρχει συνένεση των ενδιαφερόμενων μερών που να εγγυάται ότι η τεχνολογική επανάσταση συνάδει με την κοινωνική προστασία. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η ισότητα των δύο φύλων. Είναι μία από τις στοιχείες που πρέπει να εγγυηθούμε. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε μία γυναίκα να λαμβάνει χαμηλότερο μισθό από έναν άνδρα κάποια δεσμευτικά μέτρα προς ε, μεγαλύτερη διαφάνεια στο μισθολογικό μπορεί να είναι θετικά για να μπορούσουμε να κλείσουμε το μισθολογικό χάσμα, καθώς και διάφορες πρωτοβουλίες που να ευνοούν την ε, ε, συμφιλίωση της ιδιωτικής με την επαγγελματική ζωή. Οι νέοι επίσης είναι το μέλλον της Ευρώπης και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τα επίπεδα ανεργίας να φτάνουν στο 50% σε κάποια κράτη-μέλη και δυστυχώς και στο δικό μου κράτος μέλος τα διδάγματα του παρελθόντος ε, και τα αποτελέσματα της εγγύσης για τους νέους θα πρέπει να τα έχουμε κατά νου για να μην επαναληφθεί η κατάσταση αυτή. Ένα από τα σημεία που θέλω να αναφέρω και που συμπεριλάβαμε στην προηγούμενη ε, θητεία σε πολλές εκθέσεις ε, είναι το θέμα της δημογραφικής αλλαγής. Δεν αναφέρομαι στη γύρανση του πληθυσμού αλλά στην διαδικασία της απερίμωσης ε, ε, πολλών ε, και της εγκατάλειψης πολλών γεωργικών εκτάσεων. Υπάρχουν διάφορες αιτίε, δυσκολία πρόσβαση στην υγεία, στην εκπαίδευση, δυσκολία στην πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αυτό είναι κάποια παραδείγματα. Στην Ισπανία έχουμε πρόβλημα σε πολλές περιοχές και ο κίνδυνος να μην δράσουμε εγκαίρως σημαίνει ότι θα εξαφανιστούν αυτές οι περιοχές. Για να κλείσω, να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι ανταγωνιστική μόνο αν διατηρήσει ψηλά επίπεδα απασχόληση, υγείας, εκπαίδευση και κοινωνικής συμμετοχής. Και όλα αυτά δίνοντα ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα που το χρειάζονται περισσότερο. Για να το πετύχουμε, θεωρώ ότι πρέπει να υλοποιήσουμε κάποιες ενεργεί και αποτελεσματικέ πολιτικέ που να εγγυώνται ίσες ευκαιρίε ε, βάσει της αρχής της μη εισαγωγή διακρίσεων για κάθε ηλικία. Υπό την έννοια αυτή, ο κοινωνικός πυλώνας είναι ένα στοιχείο κλειδί για τη βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης και εργασίας όλων των Ευρωπαϊκών πολιτών και αποτελεί ένα χάρτη πορείας πολύ σημαντικό καθώς ε, καθορίζει προς τα που πρέπει να κινούνται οι μελλοντικέ ευρωπαϊκές πολιτικές. Επίσης ε, θεωρώ ότι το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ θα είναι ένα βασικό μέσο για να προχωρήσουμε προς την υλοποίηση αυτών των 20 αρχών που έχουμε στον κοινωνικό πυλώνα. Θα πρέπει όμως να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να ξεπεράσουμε επιτυχώς αυτές τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Γι' αυτό εγώ συμφωνώ πλήρως με τα όσα είπε η κυρία Φοντερ Λάιεν ότι η οικονομία θα πρέπει να είναι χρήσιμη για τους ανθρώπους και ότι η απασχόληση που δημιουργείται επομένως θα πρέπει να είναι ποιοτική απασχόληση και να μην επικεντρώνεται απλώς στην ποσότητα αλλά να επιτρέπει στους εργαζομένους να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή με το σεβασμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι εδώ το Eurofound μπορεί να βοηθήσει τους κυρίους βουλευτές έτσι ώστε για να μπορέσετε να νομοθετήσετε καλύτερα και να βοηθήσετε τους Ευρωπαίους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Φοντανιέ για την ε, παρουσίασή σας ε, και τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε με τον κύριο Βλάντ Μίξικ ελπίζω να το πρόφερα σωστά. Μίξιτς. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Τα ε, ονόματα στα ρουμανικά συνήθως δεν το συνηθίζουν να είναι τόσο πολύπλοκα. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να ε, ε παρευρεθώ εδώ ως υποψήφιος ε, εμπειρογνώμονας ε, για τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία και τώρα θα συνεχίσω στα ρουμάνικα. Πολλοί από όσους ε, βρίσκονται εδώ, εμού συμπεριλαμβανομένου, περνάμε περισσότερο χρόνο στο γραφείο παρά στο σπίτι μας, με την οικογένειά μας. Εγώ δυστυχώς είμαι πολύ καλή περίπτωση μελέτη γι' αυτό, γιατί η σύζυγός μου θα προτιμούσε να μην ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά δυστυχώς, δυστυχώς έχει συνηθίσει από τότε που σπούδαζα ιατρική. Γιατί σπούδασα ιατρική σε ένα μεγάλο πανεπιστήμιο στην Δυτική Ρουμανία και κατόπιν ε, μετά από 20 χρόνια άρχισα να εργάζομαι σε ένα νοσοκομείο μεγάλο με πάρα πολύ κόσμο αλλά πολύ χαμηλό προϋπολογισμό με πάρα πολλές ελλείψεις και για τους ασθενείς και για τους γιατρούς με πάρα πολύ άγχος για όλο το ιατρικό προσωπικό εκεί και μετά από κάποια χρόνια συνθετοποίησα ότι το σύστημα χρειαζόταν θεραπεία περισσότερο από τους ασθενείς και διέκοψα την ιατρική μου πρακτική και επέστρεψα στα Θρανία, στο London School of Economics, στο Λονδίνο, όπου σπούδασα πολιτικές υγείας και κοινωνικές πολιτικές. Και από τότε έχω εργαστεί στον τομέα αυτό. Σε πάνω από 7 χώρες έχω συνεργαστεί με διάφορους οργανισμούς και υπουργεία, ε, πολλές φορές ε, σε εκτελεστικές θέσεις, ενώ όλες φορές ως ε, σύμβουλος είτε για διεθνείς οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Τρέπεση, όπως το ECDC, το Κέντρο για την Πρόληψη των Νόσων εδώ στην Ευρώπη. Έπρεπε να διαμεσολαβήσω μεταξύ διάφορων φορέων με διαφορετικά συμφέροντα Πολλές ε, φορές ε, τα κατάφερα, ενώ κάποιες άλλες φορές απέτυχα και η αδράνεια των συστημάτων νίκησε. Αλλά κάθε φορά το έκανα αυτό μαζί με μια ομάδα, μαζί με άλλους και ξέρουμε όλοι σήμερα ότι πολύ περισσότερο στις πολιτικές υγείας και στις κοινωνικές πολιτικές ότι είναι αδύνατο ένας μόνος του να τα καταφέρει. Έτσι λοιπόν, αυτή η φιλοσοφία βρίσκεται και στη βάση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφαλή και την Υγεία στην Εργασία. Πρόκειται για μία από τις θεμελιώδεις αρχές του ΙΓΙΟΣΑ, ένα από τα ισχυρά σημεία του οργανισμού και ταυτόχρονα ένα από τα ευάλωτα στοιχεία Ουσιαστικά σήμερα με τον τρόπο που λειτουργεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός η Γιόσα δεν έχει συχνή επαφή με τους ε, ε, υπαλλήλους ε, αλλά έχει εθνικά στοιχεία επαφής, συνεργάζεται με τα συνδικάτα και συνεργάζεται με αυτό το δίκτυο για να συλλέξει και να παράξει όλες τις πληροφορίες, όλα τα εργαλεία που παράγει και κατά κάποιο τρόπο είναι και λογικό. Ε, είναι μικρός οργανισμός, ε, είναι ο προϋπολογισμός είναι 15,5 εκατομμύρια ευρώ, 67 εργαζόμενοι και πρέπει να ε, υπάρξει πολλή δουλειά στον οργανισμό αυτό για να είναι αποτελεσματικός. Αυτό μπορεί να είναι ισχυρό σημείο, αλλά μπορεί να είναι και ένα ευάλωτο σημείο όσο και απαραίτητα είναι τα εργαλεία που παράγονται από τον αυτός, αυτά θα έχουν πραγματικό αντικτυπώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο μόνο εκεί που έχουμε ενεργά δίκτυα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που τονίστηκε σε πρόσφατη αξιολόγηση του Γιώσα, όπου διαπιστώνεται ότι ο αντίκτυπο ε, του οργανισμού περιορίζεται από μειωμένη προβολή στα κρατη και από το γεγονό ότι κάποια εθνικά εστιακά σημεία δεν είναι πολύ ενεργά στη διάδοση των πληροφοριών η βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ του ΙΟΣΑ και των εθνικών εστιακών σημείων μπορεί να είναι κάτι χρήσιμο για να υπερβληθεί το εμπόδιο αυτό. Και μία συνεργασία ενεργή θα μπορούσε να στείλει αυτό το μήνυμα και στους τόπους εργασίας, ε, αλλά να στείλουμε και το μήνυμα ότι πρέπει να έχουμε και πρόληψη ε, στα των προβλημάτων υγεία στο χώρο εργασία. Αυτό μπορεί να είναι κάτι πολύ χρήσιμο. Αυτό είναι ε, χάρη στο πλαίσιο. Το πλαίσιο δεν είναι και ιδιαίτερα ρόδινο. Η οικονομική ύφεση, σε πολλά ουσιαστικά μειώνει τα κονδύλια που δίνονται για την ασφαλεία και την υγεία στην εργασία και δεν είναι βέβαιο ότι θα επιστρέψουν τα κονδύλια σε προκρίσεις επίπεδα. Αυτό έγινε και στο επίπεδο UOSA. Έχει παγώσει ο προπολογισμό για 4 συνεπτά έτη. Όμω παρόλα αυτά ο οργανισμό κατόρθωσε να υλοποιήσει του στόχου του. Ποιο ε, είναι τώρα το φόντο ε, στο οποίο έγινε όλη αυτή η μείωση του προπολογισμού. Να σας αναφέρω κάποια νούμερα. 4 ε, εκατομμύρια έτη ζωή χάνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω ατυχημάτων ή ασθενειών στην αγορά εργασία. 3,7 εκατομμύρια έτη ε, βιώνουν οι άνθρωποι με αναπηρίε διατροφών. Έχουμε καρκίνου, μειοσκελετικέ παθήσει, παθήσει του κυκλοφορικού. Ε, βλέπουμε ότι είναι οι περισσότερες νόσοι στους χώρους εργασίας. Έχουμε όμως μειώσει σημαντικά τα ατυχήματα σε ό,τι αφορά τη θνησιμότητα ε, έχουμε, για λόγους εργασίας. Έχουμε πολύ θλιβερά νούμερα. 52% των θανάτων προκαλούνται από καρκίνους και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ειδική περίπτωση σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Ευρώπη ο συνολικός αριθμός των ατόμων που πεθαίνουν λόγω κάποιας μορφής καρκίνου που ε, προκαλείται λόγω κάποιας έκθεσης στην εργασία είναι 80.000 ε, ετησίως και κάθε ένας από αυτούς τους θανάτους μπορεί να προληφθεί. Ο καθένας από αυτούς τους θανάτους. Το κόστος ε, είναι ανάλογο. Ε, έχουμε απώλεια σε ό,τι αφορά την παραγωγικότητα και δαπάνες στον τομέα της υγείας και μιλάμε για 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και αυτή είναι συντηρητική εκτίμηση. Αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί ο Γιώσα και δεδομένης ε, της κατάστασης και των ορίων των υφιστάμενων πόρων είναι πάλι πολύ σημαντικό να τίθενται στόχοι στη δραστηριότητα του οργανισμού. Τίθεται από το πολιετές στρατηγικό πρόγραμμα, από το Συμβούλιο και από προγραμματικά έγγραφα. Και μέχρι την έγκριση του νέου κανονισμού στις αρχές αυτού του έτους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν το στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και δεν μπορούσε να υπάρχει μια αλληλεπίδραση σε αυτή τη σημαντική φάση της θέσπισης των στόχων. Να που και αυτή η πτυχή όμως βελτιώθηκε και θα στείλει η Επιτροπή Επασχόλησης ε, έναν εμπειρογνώμονα χωρίς δικαίωμα ψήφου στο Διοικητικό Συμβούλιο, όμως αυτός ο εμπειρογνώμονας θα μπορεί να παίξει ένα ρόλο διαβίβασης μεταξύ του Τριμερούς Συμβουλίου του ΓΙΟΣΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όμως η ύπαρξη ενός εκπροσώπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο του ΙΟΣΕ έχει και μια συγκεκριμένη αξία πέρα από αυτή τη λειτουργική αξία. Βρισκόμαστε στο μέσο της τέταρτης τεχνολογικής επανάστασης, βιομηχανικής επανάστασης και ο τομέας της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία περνά από μια μεγάλη πρόκληση ο τρόπος με τον οποίο εργαζόμαστε και αλληλεπιδρούμε με τους υπαλλήλους, η ηλικία που παίρνουμε στην ταξιδότηση, όλα αυτά είναι σε πλήρη τροποποίηση και έχουμε πολλές κατηγορίες πολιτών που δεν εκπροσωπούνται ούτε από τα συνδικάτα ούτε από άλλες οργανώσεις. Μέχρι σήμερα η φωνή τους ε, δεν έχει εκπροσωπηθεί στο Συμβούλιο του ΙΟΣ, αλλά από φέτος ελπίζω και είμαι σίγουρος ότι με τη δική σας υποστήριξη και βοήθεια αυτό θα μπορέσει να βελτιωθεί. Εσείς είστε αυτοί που έχετε την πιο άμεση σχέση με τους Ευρωπαίους πολίτες και πιστεύω ότι αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία προκειμένου να τεθεί φως, να διαφωτίσουμε και τις ανάγκες υγείας των εργαζομένων. Τώρα θέλω να αναφερθώ και σε κάποιες προκλήσεις βραχυπρόθεσμα. Οι προτεραιότητες στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία δεν ε, καθορίζονται πέρα από το 2020. Πιθανότατα αυτό θα είναι ένα σημαντικό θέμα στην ημερησία διάταξη. Επίσης, όσα πρόσφατα έχει εκδώσει το πολιτεστρικό πλαίσιο μέχρι το 2023. Όμως δυστυχώ λείπει ο προϋπολογισμός. Το πολιτεστρικό πλαίσιο ίσως ένα μέρος αυτών των στρατηγικών στόχων θα πρέπει να ε, οριστούν εκ νέου προσπάθησα σε αυτό το πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να σας παρουσιάσω μόνο κάποια από τα ισχυρά σημεία και τις ευπάθειες του οργανισμού και είμαι σίγουρος ότι με τη συμμετοχή στο Συμβούλιο του ΓΙΟΣΑ ε, τόσο με την ε, ανταλλαγή πληροφοριών θα αυξηθεί και η διάδραση η δική σας μαζί τους. Θέλουμε να έχουμε ουσιαστικά ένα βλίευλο διαβίβασης ε, προκειμένου να τονίσουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη εκπροσώπηση αυτών των ομάδων όπου βασίζεται ο υγιός. Αυτό δεν είναι λεπτομέρεια, αλλά είναι σημαντικό στοιχείο για την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών. Γιατί? Η εμπειρία που έχω τα 15 χρόνια μου έδειξε ότι καμία πολιτική ε, ουσιαστικά δεν ισχύει παρά η αλήθεια. Η υγεία αποτελεί τον πλούτο μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την ομιλία σας και τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε με τον κύριο Γιάνν Κρέιμας. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλοι, ευρωβουλευτές, με μεγάλη μου χαρά αποδέχθηκα την υποψηφιότητα για την οποία θα πρέπει να λάβετε μια απόφαση απόψε το απόγευμα και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα τώρα να κάνω μια σύντομη δήλωση για εμένα καθώς επίσης και για τις ε, προκλήσεις ε, που αντιμετωπίζουμε με την ε, νέα αρχή, Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας. Ήμουνα, ε, επισκέφθηκα το Κοινοβούλιο αρκετές φορές τους τελευταίους 12 ε, μήνες ε, για να σας παρουσιάσουμε διάφορες εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις σχετικά με την εισαγωγή της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας. Αρχικά κάποια πράγματα για μένα άρχισα να εργάζομαι στον τομέα της εργασιακής κινητικότητας στην Ευρώπη πριν από περίπου 30 χρόνια. Είμαι κοινωνιολόγος ε, για ζητήματα εργασίας και ασχολούμαι με, τη, το εργασιακό δίκαιο και τις ευρωπαϊκές πολιτικές στον τομέα της εργασίας. Για ποιο λόγο αναφέρομαι τώρα σε αυτήν την περίοδο. Εργαζο... Ε, συζητήσαμε ε, για το ε, εργασιακό δίκαιο το οποίο συνδεόταν ε, με μια ε, λευκή βίβλο για την παράδοση της αρχιτεκτονικής όχι μονάχα της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης αλλά και της ενέργειας αγοράς. Η ελεύθερη μετακίνηση και η κινητικότητα των πολιτών ήδη αναφέρονται στην συνθήκη της Ρώμης το 1957 και ήταν ε, μία από τις ε, βασικότερες ελευθερίες της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης αλλά αναφέρονται επίσης και στο σχέδιο δράσης. Τότε λοιπόν ήμασταν μόλις 12 κράτη-μέλη, ακόμα είχαμε το τείχος του Βερολίνου και η ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών ήταν ένα πολύ σημαντικό θέμα. Έχω εργαστεί πάνω σε αυτό το θέμα και ως ε, Ευρωβουλευτής ήμουν ένας από τους εισηγητές ε, γνωμοδότησης ε, για την κινητικότητα των εργαζομένων και από το 2009 και έπειτα απασχολούμε στο Ινστιτούτο του Άμστερνταμ για το εργατικό δίκαιο Κατά την ε, ακαδημαϊκή μου ε, καριέρα έχω εργαστεί ιδιαιτέρως ε, για ζητήματα που αφορούν την πολιτική αυτή. σε τομείς που αφορούν τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης, την απόσπαση εργαζομένων αξιολόγηση ενισχυμένου ελέγχου και επιβολής ε, ε, το οποίο μας απασχόλησε τα τελευταία χρόνια και επίσης ως εξωτερικός εμπειρογνώμονας ε, έχω ασχοληθεί και στο πρόγραμμα Eurodetachment όπου επιθεωρήσεις εργασίας από 16 συνολικά χώρες προσπαθούν να συνεργαστούν σε εθελοντική βάση πάνω σε ζητήματα έρευνας, σχετικά με το πώς είναι δυνατόν να συνεργαστούν σε ε, υπερθυνικό επίπεδο όπου ε, υπάρχουν διαφορετικά, ε, διαφορετικές συνθήκες εργασίας σαν κράτος μέλος. αν υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας δεν είναι πάντοτε τόσο εύκολο να εντοπιστεί η ε, αρμόδια ε, αρχή, η οποία είναι υπεύθυνη σε άλλο κράτος ε, μέλος. Και έτσι λοιπόν και αυτή η εμπειρία ήταν ιδιαίτερα σημαντική για το έργο των εισηγητών κατά τα τελευταία χρόνια, οι οποίοι εργάζονταν πάνω σε ζητήματα τα οποία αφορούσαν την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας. Τώρα, όσον αφορά ε, την ΕΛΑ, την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας. Μου ζητήθηκε από την Επιτροπή σας ε, να παρουσιάσω κάποια έγγραφα θέσης, όπως επίσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κάλεσε ε, ως εξωτερικό εμπειρογνώμονα σε μια συμβουλευτική ομάδα που λειτουργεί εκεί από πέρσι το χειμώνα. Το έργο το οποίο λοιπόν έχει γίνει εκεί είναι σημαντικό ε, διότι αποτελεί μια βάση για, το, για την ε, εργασία την οποία θα αναλάβει η ε, ΕΛΑ. Τώρα η εφαρμογή όμως είναι ένα εντελώς διαφορετικό ζήτημα και σε αυτό το θέμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ε, ε, ε, εκφράζει το πνεύμα της νομοθεσίας και το οποίο στη συνέχεια, όμως στη συνέχεια η εφαρμογή της νομοθεσίας είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Έτσι λοιπόν υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις. Το έργο της ε, ELA ε, θα πρέπει να επικεντρωθεί στην βελτίωση της ε, συνεργασίας των εθνικών αρμόδιων αρχών και αυτά ήταν ένα από τα θέματα τα οποία εκφράστηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι δηλαδή το θέμα δεν είναι τόσο το να υπάρξει μια, ένας ευρωπαϊκός έλεγχος αλλά να βοηθήσει τους συναδέλφους οι οποίοι κάνουν το έργο αυτό κατά τόπους να έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται και ε, στο πρόγραμμα ε, Eurodetachment, ε, το, στο οποίο εργάστηκα όπως ανέφερα, είδαμε κάποιες πολύ σημαντικές εξελίξεις και συνεργασίες μεταξύ των Ισπανών και Γάλλων επιθεωρητών εργασίας Και επίσης έχουμε το θέμα της αποστολής ε, επιθεωρητών. Μία χώρα μπορεί πολύ εύκολα να στείλει, μπορεί και στη συνέχεια να ε, λάβει ε, ειδικού ε, στον τομέα. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε το ζήτημα της ε, κινητικότητας εργασίας ε, εργαζομένων, διότι αυτό επηρεάζει ιδιαίτερως και τις δύο χώρες. Έκανε ένα σημαντικό έργο με ανθρωπολόγους στο Πανεπιστήμιο του Πόρτο, οι οποίοι έκαναν μια ερεύνα στην Πορτογαλία σχετικά με τις συνέπειες της κινητικότητας και το 40% της, ε, του πληθυσμού της περιοχής ε, βρισκόταν ε, στο εξωτερικό, οπότε μπορείτε να καταλάβετε το πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τις αγροτικές περιοχές και το σημαντικό ρόλο που παίζουν οι γυναίκες εκεί για να βοηθήσουν την την κοινωνία. Δεν έχω όμως ρολόι μπροστά μου, οπότε δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω. Όπως και να έχει, αυτό το οποίο εκτιμώ ιδιαίτερος στα αποτελέσματα τα οποία έλαβε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε ε, να δώσουμε μια νομική αξία στις, ε, στα αποτελέσματα των ε, κοινών υπεθεωρήσεων, το οποίο ήταν σημαντικό, ένα θέμα το οποίο μας απασχολούσε από την αρχή ότι δηλαδή μπορείτε να συνεργαστείτε με τους συναδέλφους σας ε, στο εξωτερικό αλλά μπορείτε και να τους ε, επισκεφθείτε. Αυτό είναι λοιπόν ένα ε, πρώτο θέμα το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην νομοθεσία. Ένα άλλο θέμα το οποίο επίσης είναι πολύ σημαντικό είναι αρχίζουμε πολύ προσεκτικά να απομακρύνομαστε από αυτόν τον μονομερή τρόπο σκέψης, ε, απομακρυνόμαστε από τα στεγανά. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτόμαστε πιο οριζόντια, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ε, θέματα ε, με πιο οριζόντιο τρόπο και αυτό δεν είναι θέμα μονάχα συνεργασίας των διαφόρων περιφερειών που βρίσκονται κοντά μεταξύ τους, αλλά και συνεργασία μεταξύ των διαφόρων αρχών. Κλείνοντας, πιστεύω ότι το ε, Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξετάσει ε, προσεκτικά το τι θα γίνει με την ELA. Στο προήμιο αναφέρεται ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε την ε, κινητικότητα εργαζομένων και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει και μελλοντικά. Και έχω την ε, βούληση να είμαι ο δικός σας εκπρόσωπος και εκπρόσωπος της ε, Επιτροπής Απασχόλησης ε, μαζί σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε λοιπόν τις παρουσιάσεις των τεσσάρων υποψηφίων, ήταν όλες πολύ ενδιαφέρουσες. Σας ευχαριστώ πολύ και τους τέσσερις. Θα περάσουμε τώρα στις ερωτήσεις και όπως σας ανέφερα στην αρχή, ξεκινάμε με τον πρώτο γύρο με τους συντονιστές. Ξεκινάμε με τη μεγαλύτερη ομάδα, το ΕΛΚ. Η κυρία Σουίτενταλ είναι εδώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω σφυδικά. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για τις παρουσιάσεις και ε, θα ήθελα να σας συγχαρώ για τις υποψηφιότητές σας. Κύριε Μπέκερ, δεν έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν, έχω όμω ακούσει τα καλύτερα για εσάς. Και εκ μέρους του ΕΛΚ θα ήθελα να πω πως χαιρόμαστε πάρα πολύ με την υποψηφιότητά σας. Νομίζω πως ε, θα φέρετε εμπειρογνωμοσύνη στη ΣΕΔΕΦΟ. Έχω την εξή ερώτηση. Επισκέφτηκα πολλές επιχειρήσεις και πάντα άκουγα πως τα μαθήματα που προσφέρονται στους ανέργους ε, δεν χρησιμεύουν διότι δεν αντιστοιχούν στις ανάγκες αγοράς-εργασίας, σύμφωνα με τις αναλύσεις. Γι' αυτό λοιπόν ε, η ερώτησή μου είναι ε, πώς μπορούμε να αυξήσουμε το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων και να καταφέρουμε να συνδέσουμε καλύτερα τις ανάγκες των εργοδοτών με τα προσόντα των εργαζομένων και των όσων αναζητούν εργασία. Κύριε Κρέμερς, σχετικά με την ε, αγορά εργασίας και αυτά που είπατε, να σας πω πως ε, έχω ασχοληθεί στο χώρο και ήμουν αρμόδια για θέματα αγοράς εργασίας. Η δική μου εμπειρία στο εθνικό επίπεδο είναι ότι δεν υπάρχει 100% προσαρμογή ε, των συνθήκων στις πραγματικέ συνθήκες επιτόπου, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Εσείς, ε, θέλω να ρωτήσω, θα δώσετε βάση στις ιδιαίτερότητε των τοπικών κοινοτήτων, των ε, περιφερειών σε ό,τι αφορά τις ανάγκες αγορά εργασία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε λοιπόν στην επόμενη πολιτική ομάδα που έχει το λόγο. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Κυρία Γιονκέριους, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Βλέπω και νέα πρόσωπα αλλά και γνώριμα. Όλοι συνεργάζεστε λοιπόν έτσι ώστε να βελτιώσουμε την Ευρώπη και να βελτιώσουμε τα ε, εργασιακά θέματα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Αξιοπρεπούς Εργασίας, μάλιστα, και θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό να δούμε ε, και να δείτε εσείς πόσο μπορείτε να συνεισφέρετε προσωπικά σε αυτό. Μετά τις ακροάσεις των επιτρόπων, κατέστησα αφές αυτό, αλλά και το ότι η σαν πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίνει έμφαση στο, στην κοινωνική πτυχή της εσωτερικής αγοράς εργασίας της Ένωσης. Η ερώτησή μου λοιπόν για όλους έχει ως εξής. Η κυρία Φόντερ Λάιεν έχει αναθέσει στον αρμόδιο επίτροπο για την εργασία και κοινωνική υποθέσεις να καταρτήσει ένα σχέδιο δράσης για τον κοινωνικό πυλώνα. Είναι λοιπόν το πρώτο από τα καθήκοντα που θα αναλάβει ο Νίκολα Σμιτ. Οι δικές σας υπηρεσίες πώς μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτό το σχέδιο δράσης ίσως ε, μέσω της κατάρτισής του ή της ε, επεξεργασίας με προτάσεις, είτε αυτές έχουν να κάνουν με την ε, υγεία στην εργασία, είτε με την ε, κινητικότητα των εργαζομένων. Νομίζω πως όλες οι υπηρεσίες πρέπει να συνεισφέρουν σε αυτό το σχέδιο δράσης. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, εάν είναι δυνατόν εσείς, εκ μέρους της δικής μας Επιτροπής, θα έχετε τη δυνατότητα να ελέγχετε το τι κάνουν οι υπηρεσίες προς όφελος του κοινωνικού πυλώνα. Επίσης, δεν ξέρω αν αυτή η ερώτηση αρμόζει περισσότερο σε μια συνεδρία των συντονιστών, αλλά αναρωτιέμαι αν στο μέλλον θα μπορέσουν να έρθουν οι διευθυντές των Ευρωπαϊκών Αυτών Υπηρεσιών στην Επιτροπή μας. Αν θα δεχθούν λοιπόν την πρόσκληση της Επιτροπής Απασχόλησης για να έρθουν σε αυτές τις ακροάσεις και να ακούσουν και τη δική σας πλευρά. Ορισμένες υπηρεσίες είναι ενεργές εδώ και χρόνια και έχουν ήδη εδραιώσει τον τρόπο εργασίας τους. Έχουμε και μια νέα υπηρεσία. Γι' αυτό λοιπόν εγώ προσωπικά θα ήθελα πολύ να σας ε, δω μαζί με τους διευθυντέ σας. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίσουμε με την ομάδα Renew και ο κύριος Πισλάρου έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Έχω μια σύντομη ερώτηση για κάθε έναν από τους τέσσερις ομιλητές θα ξεκινήσω με το Σέντεφο. Μία από τις πραγματικότητες σήμερα είναι ότι αν και υπογραμμίζουμε τη σημασία της επαγγελματικής κατάρτισης, υπάρχει ένα στίγμα ότι οι άνθρωποι που ακολουθούν τεχνική κατάρτιση δεν είναι υπαρκώς ικανοί για άλλες σπουδές υπήρχαν, είχαν γραφτεί πάρα πολλά για την ανάγκη να υπάρχει ένα θεωρητικό σκέλος στην επαγγελματική κατάρτιση έτσι ώστε να προετοιμαστούμε για τα προσόντα του αύριο. Τώρα λοιπόν απλώς αν έχουμε την επαγγελματική οδό για όσους δεν πετυχαίνουν στη θεωρητική οδό ε, ουσιαστικά αντιμετωπίζουμε την εξής ε, πραγματικότητα ότι ε, τα προσόντα δεν ανταποκρίνονται σε ανάγκες της αγοράς. Θα πρέπει λοιπόν να μας πείτε πώς ε, θα μπορούσαμε να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα. Η δεύτερη ερώτηση είναι για την κυρία Λόπε Φοντανιέ. Στο ευρωπαϊκό εξάμεινο, εδώ και κάποιο καιρό, βλέπουμε πόσο σημαντικός είναι ο κοινωνικός διάλογος. Η ενδυνάμιση του κοινωνικού διαλόγου είναι κάτι που θα πρέπει να προωθήσουμε. Σήμερα, συνάντησα τον υποψήφιο επίτροπο, τον κύριο Ντομπρόφσκης, και είπε ότι ο κοινωνικός διάλογος είναι μία από τις προτεραιότητάς του. Το Eurofound αντικατοπτρίζει με τον καλύτερο τρόπο τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου και νομίζω ότι όλη η δουλειά που γίνεται εκεί είναι πολύ σημαντική γιατί πηγάζει από την επίδραση των εταίρων. Ε, θα ήθελα να μου πείτε ε, πώς εσείς σκοπεύετε να υποπτεύσετε αυτές τις διαδικασίες. Κύριε Κάμερς, ε, είναι κάτι καινούριο. Ένας νέος οργανισμός, η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας. Και χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω προσωπικά γιατί έχετε παίξει ζωτικό ρόλο στον πρώτο συντονισμό των συστημάτων ε, κοινωνικής ασφάλισης. Πώς βλέπετε τη σημασία της Ευρωπαϊκής Αρχής ε, Εργασίας και την εντολή που έχει για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Ε, και τέλος, η ερώτηση σε εσάς κύριε Μίξιξ. Μπορείτε να τελειώσετε παρακαλώ. Ναι, συγγνώμη. Πρέπει να είμαι δική. Λοιπόν, αν θέλετε να κατανομάσετε ένα πράγμα, ποιο θα ήταν. Συγγνώμη, πρέπει να είμαι δική. Για τους ε, πράσινους ε, θα ε, θέσω εγώ το ερώτημα. Το ερώτημα μου προς όλους τους υποψηφίους είναι πώς θα ενισχύσετε τις σχέσεις σας με τους ευρωβουλευτές και τι είναι αυτό που σας καθιστά ιδανικούς για, αυτήν, για, την εκάστοτε, για τον εκάστοτε οργανισμό. Και συνεχίζουμε με το ID. Δεν βλέπω. ECR. Δεν είναι. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Συγχαρητήρια ε, σε όλους τους ε, υποψηφίους για τις υποψηφιότητες τους και θα επαναλάβω μία ερώτηση που ήδη τέθηκε. Ε, πώς ακριβώς ε, σκοπεύετε να συνεργαστείτε με την Επιτροπή μας, ε, πόσο συχνά θα συζητάτε και θα έρχεστε σε επαφή μαζί μας και για την υποψήφια του Eurofound ποια ε, ε, θέσεις σας ε, για τις προκλήσεις της αγοράς εργασίας. Έχουμε μια γυράσκουσα κοινωνία, οπότε τι πιστεύετε μπορούμε να κάνουμε ούτω ώστε να βελτιωθούν οι δεξιότητες των ηλικιωμένων εργαζομένων. Το θέμα αφορά και τις ψηφιακές δεξιότητες αυτής της ομάδας. Στον κύριο Μπέκερ τώρα, ε, πώς, μπορούμε καλύτερα να συνεργαστούμε με τους επιχειρηματίες ε, ε, για το θέμα της απασχόλησης και της κατάρτισης για τον κύριο Βλάντ Μίτσιτς. Της, το θέμα αφορά την προστασία της υγείας των εργαζομένων σε γραφεία. Τι μπορεί να γίνει εκεί. και η ερώτηση για την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας, η LA, αναφέρθηκε ότι ε, κατά τη διάρκεια των εργασιών που έγιναν για, τις, ε, για την κατάρτιση των ορμοδίτων, Τη ε, της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας αναφερθήκατε στο ζήτημα των ε, κοινών ελέγχων. Όμως το πραγματικό πρόβλημα είναι η έλλειψη γνώσης ε, όπου η οι επιχειρήσεις αποσπούν νόμιμα τους εργαζομένους και όταν υπάρχει αμφιβολία για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν την έδρα τους εκεί όπου γίνεται η εργασία τότε ε, θα πρέπει η επιθεώρηση ε, της ε, η επιθεώρηση της μίας χώρας που υποδέχεται δεν έχει πρόσβαση στην επιθεώρηση εργασίας της χώρας που αποστέλει τους εργαζομένους. Οπότε, τι έχετε να πείτε για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των επιθεωρήσεων εργασίας των διαφόρων χωρών. και ε, τι έχετε να πείτε σχετικά με το πώς θα μπορεί να γίνεται η ανταλλαγή πληροφοριών. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε με την ΚΟΕ. Δεν έχουμε ερώτηση από εκεί. Και τώρα θα περάσουμε στις απαντήσεις που θα δώσουν οι υποψήφοι. Ε, τρία λεπτά ο καθένας ε, για να απαντήσουν στις ερωτήσεις αυτές και θα έλεγα να ξεκινήσουμε και πάλι με τον κύριο Μπέκα και να ακολουθήσουμε την ίδια σειρά που είχαμε και προηγουμένως. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω τώρα να απαντήσω στις ερωτήσεις που μου θέσατε σχετικά με την ερώτηση για τους ε, ε, ανέργους και τα σεμινάρια που θα προσφέρονται για αυτούς για να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Πολύ συχνά λέμε ότι λείπουν οι αναλύσεις και ακριβώς αυτό είναι ένα θέμα ε, και αναφέρεται στην εντολή της ε, ΣΕΝΤΕΦΟΠ ότι θα πρέπει να κάνει δηλαδή αναλύσεις ε, που, τις οποίες χρειάζεται η αγορά τόσο οι εργοδότες όσο και οι εργαζόμενοι και εδώ στην έκθεση αναφέρονται οι βασικές δράσεις της ΣΕΝΤΕΦΟΠ να υπάρχει μια σύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης και της αγορά εργασίας φυσικά και θα προωθήσουμε ε, κάτι τέτοιο το οποίο θα ε, παρακολουθεί την ε, δράση αυτή. Τώρα στο ερώτημα της κυρία Γιουνκέριους που συνδέεται με την Παγκόσμια ημέρα για, τις, για την αξιοπρεπή εργασία, αυτό θα βρεθεί, στο, θα εντοπιστεί στο ρόλο των κοινωνικών εταίρων. Δεν μπορώ να βρω κάποια εναλλακτική σε αυτό το θέμα. αναφερθήκατε στο όραμα της ε, κυρίας Φοντελάιερ σχετικά με τον ε, κοινωνικό πυλώνα δικαιωμάτων. Μου κάνει εντύπωση το ότι ε, καταφέραμε κάτι αυτό. Ήταν ένα πολύ σκληρό έργο. Θα εργαστούμε πάνω σε αυτό και ναι φυσικά και θα το έχω υπόψη μου κατά τις εργασίες μου. την ερώτηση του κυρίου Μπισλάρου, όντως έχουμε αναγνωρίσει το στίγμα το οποίο υπάρχει. Η επαγγελματική κατάρτιση δεν έχει ε, το ίδιο πριστής και δεν έχει και τις ίδιες απολαβές όπως ε, με την ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Η ε, ΣΕΝΤΕΦΟΠ έχει ως στόχο της ότι θα πρέπει να υπάρχει θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία ε, μεταξύ της ε, επαγγελματικής κατάρτισης και της ακαδημαϊκής ε, κατάρτισης και να μην λέμε ότι η επαγγελματική κατάρτιση στη χώρα μας είναι κατώτερη από την ακαδημαϊκή. Τώρα όσον αφορά την ε, διατήρηση της ε, σύνδεσης ε, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο για μένα θα ήθελα να το θέρω εγώ, διότι έλαβα ένα έγγραφα που λέει ότι μας καλύπτονται τα έξοδα για δύο επισκέψεις το χρόνο. Εγώ θα ήθελα να έρχομαι πιο συχνά. Ε, όμως ε, θα πρέπει να υπάρχει ε, μεγάλη συνεργασία και επαφή μεταξύ της Επιτροπής αυτής και των εμπειρογνωμόνων που αποστέλλεται. Τώρα τι είναι αυτό το οποίο με καθιστά ιδανικό είναι το γεγονός ότι για πάρα πολλά χρόνια εργαζόμενο στον τομέα έχω καταρτήσει ε, γνωμοδοτήσεις πάνω σε αυτό. Ε, βρισκόμουν στην Επιτροπή Κούλτ η οποία επικεντρώνεται περισσότερο ε, στο θέμα της εκπαίδευσης παρά στο θέμα του ε, πολιτισμού και εκεί έχουμε ασχοληθεί με πάρα πολλά ζητήματα τα οποία αφορούν το ζήτημα της εκπαίδευσης οπότε από εκείνη την περίοδο έχω την απαραίτητη εμπειρία ε, για να αναλάβω αυτήν την θέση. Τώρα το ερώτημα σχετικά με το πώς ε, θέλω να συνεργαστώ με αυτήν εδώ την Επιτροπή και πόσο συχνά θέλω να επικοινωνώ. Ε, προσωπικά πιο συχνά από ό,τι λέει το έγγραφο το οποίο ορίζει ε, δύο φορές τον χρόνο. Γνωρίζω ότι η γραμματεία θα με ενημερώσει και θα με βοηθήσει πάνω σε αυτό τώρα σχετικά με το ποιο μοντέλο συνεργασίας θεωρώ ότι είναι το καλύτερο. Δείχνουν όλα ότι η ε, εργασία με τους, ε, συνεργασία με τους ε, κοινωνικούς εταίρους, οι κανονισμοί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στους οποίους βοήθησαν να καταρτιστούν είναι ξεκάθαρο το γεγονός ότι οι κοινωνικοί εταίροι αποτελούν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπέκα. Και συνεχίζουμε με την κυρία Φοντάνια. Τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εγώ νομίζω ότι όλες οι ερωτήσει σχετίζονται μεταξύ τους. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες. Η κυρία Γιονγκέριος μίλησε για εξωπρεπή εργασία. Αυτό που δεν μπορούμε να παραδεκτούμε είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλοί Ευρωπαίοι που είναι φτωχοί εργαζόμενοι εργάζονται, αλλά δεν μπορούν να ζήσουν από την εργασία τους. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, όταν μιλάμε για μια ποιοτική απασχόληση, αυτό πρέπει να αναζητήσουμε. Τι μπορούν να κάνουν ε, οι οργανισμοί και συγκεκριμένα το Eurofound. Θα πρέπει να εργαστούν για τα δεσμικά όργανα και συγκεκριμένα για αυτό το κοινοβούλιο. Εγώ, βάσει της ε, εμπειρίας μου, γνωρίζω ότι πολλές φορές μας λείπουν συγκεκριμένες περιπτώσεις και οι οργανισμοί μπορούν να μας δώσουν αυτά τα στοιχεία. Έχουν πιλωτικά σχέδια. Ε, επίσης, το Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει να υλοποιηθούν τέτοια πιλωτικά σχέδια. Τι θα γίνει με τις νέες θέσεις απασχόλησης ε, και τις συνέπειες. Ε, έχουμε το θέμα της ψηφιοποίησης. Φοβούνται οι εργαζόμενοι Μπορούμε να μιλήσουμε και για τους πιο ηλικιωμένου ε, εργαζομένους, οι οποίοι ε, φοβούνται ε, ενώπιον της ψηφιοποίησης, φοβούνται πως αντικατασταθούν με τα ρομπότ. Έτσι λοιπόν θα πρέπει οι οργανισμοί αυτοί να κάνουν μελέτες για να δουν πώς μπορούν να αποκτήσουν νέα προσόντα οι εργαζόμενοι για να συνεχίσουν να εργάζονται και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις επιχειρήσεις. Εγώ ξέρω ότι στο Eurofund μελετάτε ένα θέμα πολύ σημαντικό για όλους εσάς, ε, ελάχιστος μισθός όλα τα κράτη-μέλη, ο κατώτατος μισθός. Θα συνεχίσουμε τη μελέτη του θέματος αυτού. Ένα άλλο ε, θέμα είναι η εγγύηση για τα παιδιά. Εγώ νομίζω ότι οι περισσότεροι βουλευτές συμφωνούσαν με τον να μια εγγύηση για τα παιδιά. Όμως ε, γνωρίζουμε ακριβώς ε, σε τι συνίστατο. Αυτό είναι πιο πολύπλοκο. Δηλαδή αλλάζει αναχώρα, αλλά θα πρέπει και να ορίσουμε τι εννοούμε με τον όρο εγγύηση για τα παιδιά. Και ένας οργανισμός όπως το Eurofound μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ τα θεσμικά όργανα και τους βουλευτές και τα κράτη-μέλη που θα πρέπει να προβούν στην εφαρμογή, πώς μπορούν να υποστηρίξουν την εγγύηση για τα παιδιά. Και αμφισβήτητα πρέπει να μιλήσουμε και για προπολογισμό. Χρειάζονται χρήματα για αυτά τα έργα. Γι' αυτό είναι και σημαντικά τα πιλωτικά έργα. Τώρα, κύριε Πασλάρου, κοινωνικός διάλογος είναι απαραίτητος. Και βλέπουμε ότι στις χώρες όπου λειτουργεί περισσότερο κοινωνικός διάλογος, είναι πιο εύκολο για τις επιχειρήσεις να μπορέσουν να έρθουν σε συνεννόηση με τους εργαζομένους και να δημιουργήσουν αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας προκειμένου να υπάρχει ποιότητα ζωής για όλους τους εργαζομένους. Κυρία Πρόεδρε, ποιος είναι ο ρόλος μας Νομίζω ότι αυτό εσείς θα πρέπει να το προσδιορίσετε. Μπορούμε να διευρύνουμε αυτό το ρόλο, αν το επιθυμείτε. Εγώ πιστεύω ότι είναι σημαντικό. Έχουμε κάποια εμπειρία και ως πρώην βουλευτές και ξέρουμε τι βοήθεια μπορούν να προσφέρουν αυτοί οι οργανισμοί. Επίσης ξέρουμε και την προβληματική. Και εγώ νομίζω ότι θα μπορούσε να καθορίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε και θα μπορούσαμε να είμαστε η φωνή και του οργανισμού αλλά και του Κοινοβουλίου, προκειμένου να υπάρχει ένας βέλτιστος συντονισμός. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε και ο λόγος στον κύριο Μίξιτ Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε μια ερώτηση που φαίνεται ότι απευθύνεται και στους τέσσερις. Ποιος είναι ο ρόλος των εμπειρογνωμόνων στα συμβούλια των τεσσάρων οργανισμών βάσει της ε, προηγούμενης εμπειρίας μου καθώς ε, έχω εργαστεί και για οργανισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ζωτικό και ότι δεν θα χρησιμοποιήσω ένα πολύ κοινό όρο, το πόσο πελάτης ορίζει τους όρους αναφοράς και τους ρόλους. Και μάλιστα ο πελάτης είστε εσείς εδώ, τα μέλη της Επιτροπής. Επομένως, αν μιλάμε για το πώς φορές θα συναντηθούμε. Προσωπικά, Δεν ε, θα ενδιαφερόμουν να καταλάβω τη θέση αν δεν μπορούσε να επικοινωνώ μαζί σας το συχνότερο, όσο δυνατόν συχνότερα. Ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα μπορέσει να μας συμπεριλάβει και μας όσο το δυνατόν ε, με μεγαλύτερη δυναμική και να ζητά από εμά πληροφορίες και υποστήριξη για τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με τους τομείς στους οποίους απασχολούμαστε. Τώρα να περάσω στην πιο συγκεκριμένη ερώτηση της κυρίας Γιονγκέριους. Υπάρχει ένας ε, διεθνώς αποδεκτός στόχος. Είναι πολιτική και στο ευρωπαϊκό επίπεδο που μπορεί να συνοψιστεί. Υγεία σε όλους. Και όπως ξέρετε, σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η υγεία και στο εργατικό δυναμικό και η υγεία στον χώρο εργασίας βρίσκονται στις αρμοδιότητες πολλών οργανισμών. Αν δείτε τι συμβαίνει σε εθνικό επίπεδο, θα έχετε μάλλον τουλάχιστον τέσσερα υπουργεία ή οργανισμούς με πολλές επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες. Ο κοινωνικός πυλώνας είναι μία από τις καλύτερες ευκαιρίες για να προσπαθήσουμε να κάνουμε να συμμετέχουν όλοι οι υπάλληλοι που δεν εκπροσωπούνται πάντοτε ούτε ε, συμμετέχουν στις οργανώσεις εκπροσώπησης και στη τριμερή δομή τώρα η τριμερή δομή του Συμβουλίου θα πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες εξελίξεις. Γιατί όπως είπα και πριν, ε, η βιομηχανική επανάσταση θα την προκλήσει σε όλους μας. Κύριε Πεσλάρου, πολύ σύντομα θα σας απαντήσω. Τώρα, στην Ευρώπη κάποιες ε, διαταραχές που αφορούν την κατάθλιψη και ε, αποτελεί την τρίτη αιτία νόσου και περίπου το 40% των ε, αρμοδίων οργανισμών ε, μας λένε ότι δεν έχουν επαρκή στοιχεία σε σχέση με αυτές τις ε, ψυχικές νόσους. Έτσι λοιπόν αν το δούμε και από ιατρική, επιδημιολογική σκοπιά και κοινωνική σκοπιά είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πρέπει να δώσουμε πολύ μεγαλύτερη προσοχή σε αυτό το θέμα και ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφαλή και την Υγεία Συνεργασία θα μπορούσε να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Τώρα, για του εργαζομένου στα γραφεία. Μου αρέσει αυτό το θέμα. Θα πρέπει να είμαι σύντομο βέβαια, γιατί ήδη έχω υπερβεί το χρόνο. Να σας πω, παραδείγματος χάρη, τον Οκτώβριο του 2020, όσα θα ξεκινήσει τη νέα διετή εκστρατεία που στοχεύει στις μυοσκελετικές ε, παθήσεις και όπως ε, ξέρετε κυρίως πάσχουν από αυτές ε, οι εργαζόμενοι στα γραφεία. Είναι ουσιαστικά τύχη που ακριβώς ο οργανισμός θα αρχίσει να εργάζεται για αυτό το θέμα. Όμως μάλλον είναι, δεν υπήρχε και κάποια έλλειψη στα στοιχεία αυτά, γιατί αυτά τα θέματα αποφασίζονται από το Συμβούλιο τρία έτη πριν. Έτσι λοιπόν νομίζω, ή μάλλον είμαι σίγουρος ότι η Επιτροπή θα έχει σίγουρα κάτι να πει, τουλάχιστον ε, να δώσει κάποια στοιχεία στον οργανισμό σε σχέση με το ποια είναι τα πιο σημαντικά θέματα προς επιλογή. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αυτές οι διετες εκστρατείε είναι από τις πλέον ορατές, είναι ένα από τα πιο επιτυχή προϊόντα του όσου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος τώρα στον κύριο Κρέμερς για να απαντήσει στις ερωτήσεις και μετά θα περάσουμε στο δεύτερο γύρο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω κι εγώ να είμαι σύντομος. Κυρία Σουίτεντάλ, Αναφερθήκατε στις τοπικές ανάγκες και τις επιπτώσεις σε τοπικό επίπεδο. Έχω πει κατά τη διάρκεια των συζητήσεων ποια είναι η προστιθέμενη αξία που θα αποκομίσουμε αν δημιουργήσουμε ένα κεντρικό επίπεδο της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας. Αν δείτε τις διάφορες πρωτοβουλίες βάσης, τις οποίες συμμετέχουν και πάρα πολλοί Σουηδοί συνάδελφοι, θα παρατηρήσετε πως υπάρχει επίγουσα ανάγκη ανταλλαγής εμπειριών. Δηλαδή, πώς να αντιμετωπίσουμε διάφορες ε, περιπτώσεις, διάφορους τεχνητούς ε, διακανονισμούς ε, για την πρόσβαση στην αγορά, για παράδειγμα. Έχουμε δημιουργήσει την ελευθερία εγκατάσταση στην Ευρώπη, τις σχετικές υπηρεσίες, όμως τα μέσα που έχουμε για να ελέγχουν εάν γίνονται τα πράγματα σωστά ε, από κοινωνικής άποψης έχουν όρια γεωγραφικά. Οι επιθεωρήσεις εργασίας δεν μπορούν να δράσουν εκτός της ε, περιφέρειας αρμοδιότητας. Τα διάφορα, διάφοροι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης έχουν και αυτή η περιορισμένη εμβέλεια και να μην αναφερθώ στις φορολογικές αρχές, οι οποίες δεν έχουν καμία απολύτως δικαιοδοσία εκτός έδρας. Υπάρχει λοιπόν μια αυξανόμενη ανάγκη για συνεργασία και νομίζω πως η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας είναι η πρώτη υπηρεσία που θα νομιμοποιήσει τη συνεργασία αυτή. Και εδώ να απαντήσω και στον συνάδελφο που ρώτησε κάτι σχετικό, ότι Είμαι υπέρ των κοινών επιθεωρήσεων εργασία, όμως και πάλι πρέπει να εστιάσουμε εδώ στην ανταλλαγή πληροφοριών. Αυτή τη στιγμή διενεργείται μια αξιολόγηση των ιανίων σημείων επαφής και των ε, γραφείων σύνδεση. Σίγουρα μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα, παρότι Έτσι θα μεταδώσουμε και θα ανταλλάξουμε αυτές τις πληροφορίες. Ε, νομίζω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας μπορεί να αναλάβει ρόλο παρακολούθησης και από την άλλη να δώσει το μήνυμα σε αυτούς ε, τους φορείς να συνεργαστούν με τις οργανώσεις βάσης, να καταφέρουν να βελτιώσουν έτσι την κινητικότητα των ε, εργαζομένων. Και να απαντήσω και σε άλλες δύο ερωτήσεις που μου έγιναν από την κυρία Γιονγκέριους και τον κύριο Πισλάρου Όταν ο πρόεδρος Γιούνκερ έκανε λόγο για την αρχιτεκτονική δομή της ενίας αγοράς, ήταν αρκετά περίεργο το γεγονός ότι υπάρχει μεν Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, αλλά δεν υπάρχει κάποια αρχή που να ελέγχει μία από τις θεμελιώδεις ελευθερίες της Ένωσης. Και αυτό νομίζω έδωσε το μήνυμα να κοιτάξουμε ξανά την δομή της ε, ενιαίας αγοράς. Και νομίζω πως δεν μπορώ να σας προτείνω κάποια συγκεκριμένη πρωτοβουλία, αλλά αν καταφέρουμε να ενσωματώσουμε όλες τις επιτυχίες, δεν θα μπορέσουμε να εξετάσουμε με επιτυχία τα επιμέρους προβλήματα. Όλα συνδέονται μεταξύ τους. Και για να επιβιώσουν εργαζόμενοι στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας, διότι μην ξεχνάμε ότι η ελεύθερη κυκλοφορία είναι μία από τις βασικές αρχές της Ένωσης, χρειάζεται να ενσωματωθούν όλα αυτά. Και όταν συζητούσαμε για το συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης, πολύ συχνά ακούγαμε ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με την ε, κινητικότητα στην εργασία. Νομίζω πως τώρα δεν υπάρχει πια παρανόηση ή παρεξήγηση. Γνωρίζουμε ότι όταν πάει κάτι στραβά σε έναν τομέα, επηρεάζονται κι άλλοι. Και νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα, με καλέσατε και μου ζητήσατε να κάνω μια πρόταση για τον κοινωνικό πυλώνα. Να σας πω ότι στο θέμα της φορολόγησης ε, υπάρχουν ενδιαφέροντα νέα. Για παράδειγμα, αν υπάρχουν κάποιες διασυνοριακές αλυσίδες παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, Οι φορολογικές αρχές δεν τις αντιμετωπίζουν ξεχωριστά, αλλά ως ε, μία φορολογική οντότητα. Και αυτό νομίζω είναι κάτι που αξίζει να αντικατοπτριστεί και στον ε, κοινωνικό τομέα. Στη, στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας ήδη έχουν γίνει βήματα μέσω των ευρωπαϊκών υπηρεσιών, διότι, για παράδειγμα, ισχύει ότι ανεξάρτητα από το που από το από πού προέρχεται ο εργαζόμενος, η ευθύνη είναι στον, ε, στο χώρο εργασίας. Ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε τώρα στο δεύτερο γύρο ε, ερωτήσεων και θα ζορίσουν λίγο τα πράγματα. Θα ήθελα λοιπόν να επενθυμίσω ότι όσοι θέλετε να κάνετε ερωτήσεις έχετε μόνο ένα λεπτό για να το κάνετε αυτό. Και έπειτα οι προσκεκλημένοι θα έχουν μόνο δύο λεπτά χρόνο για να απαντήσουν. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να τηρήσετε το χρόνο ομιλίας, να προσπαθήσουμε τουλάχιστον. Έχω λοιπόν ένα κατάλογο μελών που έχουν ζητήσει το λόγο. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία Άννα Σαλεύσκα από την ομάδα ECR. Μετά ο κύριος Λένερτς από το ΕΛΚ, η κυρία Άννα Σαντέρ από το ΕΛΚ, Κυρία Τρία Λενουά από το Renew. Ο κύριος Πάτον. Και τέλος, εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο κύριος Ντάνιελσον. Έχω ξεχάσει κάποιον μήπως? Όχι. Ξεκινάμε με την κυρία Ζαλεύσκα. Έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Συγχαρητήρια σε όλους τους προσκεκλημένους. Μία ερώτηση για τον κύριο Μπέκερ. Βλέπουμε, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι το σύστημα δύο κατευθύνσεων στην εκπαίδευση είναι η λύση για το μέλλον. Πολλές χώρες έχουν εισαγάγει το σύστημα αυτό, πολλές ήδη το χρησιμοποιούν, υπάρχει διαδίκτυο σε όλα τα σχολεία, είναι πάρα πολύ σημαντική να πω εδώ η πρόσβαση στο διαδίκτυο στα σχολεία. και μπορούμε να το παρουσιάσουμε μάλιστα ακόμα καλύτερα στο πλαίσιο της, της εκπαίδευσης δύο κατευθύνσεων. Εσείς έχετε κάποια ιδέα για το πλαίσιο το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Ίσως το Ευρώπη 2020 να ήταν μια καλή ιδέα και αναφέρομαι στην γενική εκπαίδευση και όχι στην επαγγελματική. Πώς λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω, μπορούμε να αναλύσουμε την ποιότητα της άτυπης εκπαίδευσης ε, μέσω, για παράδειγμα, διαδικτυακών μαθημάτων οι αξιολογήσεις ε, δεν αναφέρονται πάντα στην ποιότητα και πώς μπορούμε εσωτερικά να αξιολογήσουμε την ποιότητα της εκπαίδευσης. Αυτά και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριος Λένας Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πολύ που βρίσκεστε εδώ, εσείς οι τέσσερις υποψήφοι, είστε γνώριμα πρόσωπα. Χαίρομαι πολύ λοιπόν που σας βλέπω. Μία ερώτηση για όλους. Άκουσα αρκετά για το ρόλο σας ως ε, η φωνή του Κοινοβουλίου, ως εκπρόσωπου της Επιτροπής. Από την άλλη, ο κανονισμός αναφέρεται με σαφήνεια σε ένα ανεξάρτητο σώμα που θα διοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς λοιπόν πώς ε, θα μπορέσετε να ισορροπήσετε μεταξύ αυτής της ανεξαρτησίας και αυτών που έχετε πει. Έπειτα, είμαι... παρακολουθώ πολύ, από πολύ κοντά την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας. Εσείς Πού μπορείτε να βοηθήσετε περισσότερο στην εφαρμογή του κανονισμού, θεωρείτε. Έπειτα, η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασία είναι μια καινούργια υπηρεσία. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει την ερχόμενη εβδομάδα για πρώτη φορά. Πώ λοιπόν εσεί μπορείτε να διασφαλίσετε ότι οι εμπειρογνώμονε θα είναι παρόντε την ερχόμενη εβδομάδα για την πρώτη αυτή συνεδρίαση. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με την κυρία Ζάντα. Ευχαριστώ. Εγώ δεν έχω ερώτηση. Αυτό θα μας επιτρέψει να κερδίσουμε χρόνο σε απαντήσεις. Απλώς ένα σχόλιο θέλω να κάνω. Να πω ότι χαίρομαι που βλέπω τους τέσσερις εμπειρογνώμονες σήμερα εδώ ενώπιόν μας. Δύο τους γνωρίζω ήδη, γιατί μαζί αγωνιστήκαμε. Και εγώ μάλιστα ήμουν εισηγήτρια για την αναθεώρηση του κανονισμού σε αγωνιστήκαμε έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορεί να κάνει τη φωνή του να ακουστεί και η φωνή του Κοινοβουλίου εκφράζεται μέσω ημών σήμερα και μάλιστα το ίδιο και τους επόμενους μήνες. Θα ήθελα λοιπόν ε, να ε, σας πω καλό κουράγιο ότι έχετε πολύ μεγάλη ευθύνη καθώς είστε οι πρώτοι εμπειρογνώμονες ε, που θα εκπροσωπήσουν το Κοινοβούλιο σε θέματα πραγματικά ουσιώδη και που είναι πολύ σημαντικά για μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η κυρία Τριέλη Νουάρ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω γαλλικά. Κύριε Μίξιτς, κύριε Λοπεφαντανιέ, στις αντίστοιχες διαδρομές σας διαπιστώσατε τις ε, μεγάλες αρισότητες ε, μεταξύ των πολιτών σε ό,τι αφορά την υγεία σας. κύριε Μίξιτς. Συγκρίνατε τα συστήματα, τα υγειονομικά μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης ε, και κύριε Λοπεφτανιέ, επειδή ήσασταν στην ομάδα την διακομματική για την καταπολέμηση της ανέχειας στο Κοινοβούλιο. Ξέρετε, το προσδόκιμο ζωής μπορεί να διαφέρει μέχρι και 8 έτη ανάλογα με το κοινωνικό και οικονομικό στάτους των πολιτών, ανάλογα με τα επίπεδα του εισοδήματός τους και το μορφωτικό τους επίπεδο και φυσικά ανάλογα και με την εργασία της απουσίας εργασίας, ανάλογα με το μισθό, τον τρόπο ένταξης ή επανένταξης και ανάλογα με τις συνδίκες υγείας, ε, όλα αυτά είναι καθοριστικά. Και σας ευχαριστώ που υπενθυμίσατε τον αριθμό των καρκίνων που μπορούμε να αποφύγουμε χάρη σε φιλόδοξες πολιτικές πρόληψης ε, στην εργασία. Πώς ε, εσείς ε, θεωρείτε ότι θα ελαιοποιηθεί ο ρόλος των οργανισμών ε, για να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες στον τομέα της υγείας. Ευχαριστώ. Και συνεχίζουμε με τον κύριο Πάτν. Ευχαριστώ πολύ. Έχω μία ερώτηση για τον κύριο Μπέκα. Έχετε επιλεγεί ως εμπειρογνώμονος για τη ΣΕΔΕΦΑΠ, όμως από την ε, παρουσίασή σας δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η εμπειρογνωμοσύνη σας. Ε, έχετε εργαστεί στις κοινωνικές ασφαλίσεις, συντάξεις, ε, στον τομέα της διαφήμισης, όμως δεν είπατε απολύτως τίποτα σχετικά με την ε, επαγγελματική κατάρτιση, την έρευνα στους τομείς, ε, τα προβλήματα σχετικά με την αναγνώριση προπτυχίων, αλλά ε, και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι που ζουν σε απόκεντρε περιοχέ. Και αναρωτιέμαι λοιπόν αν γνωρίζετε πόσοι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν κάποια κατάρτιση, πόσοι νέοι εγκαταλείπουν το σχολείο χωρί καμία κατάρτιση. Αναρωτιέμαι αν γνωρίζετε πόσε θέσει πρακτική υπάρχουν στην ίδια σα τη χώρα χώρα. Με όλο το σεβασμό, λόγω της ε, έλλειψης εμπειρίας στον τομέα, εσείς είστε ο μαθητευόμενος, ε, οπότε θα δίνατε στον εαυτό σας αυτήν την ε, δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Και στον τελευταίο ομιλητή, ο κύριος Τάνιεσον από το S&D. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τις παρουσιάσεις. Έχω μία ερώτηση για τον κύριο Κρέμερς. Ο κανονισμός της ELA λέει ότι τα συνδικάτα και ε, οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν ε, να θέσουν υποθέσεις σε εσάς ποιος, ε, ποιο, με ποιο τρόπο λοιπόν θα λύσετε τα ε, προβλήματα αυτά. Για παράδειγμα ένα συνδικάτο σας καταγγέλει ότι υπάρχει μια επιχείρηση η οποία πληρώνει λιγότερο από τα συμφωνηθέντα. Πώς ακριβώς θα το κάνετε, θα επιλύσετε αυτές τις διαφορές όταν υπάρχει διασυνοριακή διάσταση. Οι Σουηδικές αρχές κάνανε πρόσφατα σε κατασκευαστικές εταιρείες, το 25% έκλεισε αμέσως λόγω παρατυπιών. Ε, η ΕΛΑ θέλει να κάνει ε, αλλαγή, να, κάνει, ε, να βοηθήσει από τώρα ή θα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές ούτως ώστε να μπορεί να παρέμβει. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ κλείνει ο γύρος των ερωτήσεων και τώρα θα περάσουμε πάλι στις απαντήσεις. Κάθε υποψήφιος έχει δύο λεπτά και θα ξεκινήσουμε πάλι με τον κύριο Μπέκερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να δώσω την απάντηση στον ε, ε, στην κυρία Ζελεύσκα όσον αφορά την αναγνώριση των αποφύτων διπλής κατάρτισης υπάρχουν ακόμα χώρες ε, όπου δεν έχει επιτευχθεί το επίπεδο που θέλουμε. Σε Αυστρία και Γερμανία το επίπεδο είναι πολύ ανεβασμένο όμως σε όλη την Ευρώπη θα πρέπει να εργαστούμε ούτως ώστε επιτέλους ε, μία μη ακαδημαϊκή πορεία ε, κατάρτιση να έχει και αυτή την απαραίτητη αξία στην αγορά ε, εργασίας και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει επιληθεί ακόμα. Τώρα η ικανότητα απασχόλησης δεν είναι παράγοντα σχετικά με το πώς θα αξιολογούμε την κατάρτιση. Είναι ένας δρόμος προς την απασχόληση ή ε, είναι μια κατάρτιση ιδεών. Νομίζω ότι η ικανότητα να απασχοληθεί κανείς είναι αυτό το οποίο θα μας απασχολεί. Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες ε, πάντοτε ε, βρίσκονται στη διάθεση αυτών που τους αποστέλουν και για αυτούς για τους οποίους εργάζονται Πιστεύω λοιπόν ότι εφόσον ναι, δεν υπάρχουν εμπειρίες θα πρέπει να μείνουμε ανοιχτοί, θα πρέπει να αξιολογούμαστε και έτσι λοιπόν και από αυτήν εδώ την Επιτροπή θα παρακολουθούμαστε και ταυτόχρονα ε, και από τον εκτελεστικό διευθυντή θα ε, ελεγχόμαστε. Όλοι μας ε, θα πρέπει να είμαστε ανεξάρτητοι και πιστεύω ότι και θα το καταφέρουμε. Τώρα σχετικά με το πώς Ε, αξιολογώ το ζήτημα της CLA διότι ήμουν επικριτικός απέναντί της ε, είναι ένα ε, θέμα το οποίο μας αποσχολεί ιδιαίτερος τώρα το πώς θα με επηρεάσει αυτό στο έργο μου, στο έργο μου στη ΣΕΝΤΕΦΟΠ είναι το γεγονός ότι και πάλι η αγορά εργασίας βρίσκεται στη διάθεση μιας, ενός οργανισμού που έχει την εμπειρία και την γνώση για να χειριστεί το θέμα αυτό. Τώρα κυρία Νουάγα αναφερθήκατε στο ζήτημα του καρκίνου, δεν είμαι ειδικό πάνω στο θέμα, όμως ε, πιστεύω ότι αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό ε, πρόγραμμα το οποίο το ζητούσαμε πάντοτε. Πάντοτε θέλαμε ένα μεγάλο πρόγραμμα να θέσουμε ε, ένα νέο στόχο που είναι η εξάλληψη του καρκίνου στο άμεσο μέλλον. Κύριε Πέτεν, ε, η δική μου κατάρτιση είναι αυτή που σχετίζεται με το ότι δεν σπούδασα ε, για το θέμα της αγοράς εργασίας ε, αλλά ήμουν εισηγητής για το ζήτημα της δυτής κατάρτισης της επαγγελματικής κατάρτισης. Επίσης ήμουν επιχειρηματίας, είχα προσλάβει κόσμο και εδώ στο κοινοβούλιο επίσης απέκτησα πολύ σημαντική γνώση για αυτό το θέμα όπως ε, για παράδειγμα όταν βοήθησα στην ε, κατάρτιση του ε, Ευρωπαϊκού Δικτύου για την κατάρτιση και για αυτό τον λόγο Ε, θα εργαστώ ιδιαιτέρως ε, για την ε, πρόσβαση που θα έχουν οι νέοι από απόκεντρες περιοχές στην αγορά εργασία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπέκερ και συνεχίζουμε με την κυρία Φωτανία παρακαλώ. Θα είμαι σύντομη πρόεδρε. Γιατί πιστεύω ότι ο σύντροφος Μπέκερ απάντησε και κάλυψε τις κοινέ ερωτήσεις. Κύριε Λένερ, είναι παλιό συντροφό μου. Πώς μπορούμε να είμαστε ανεξάρτητοι και ταυτόχρονα να εκπροσωπούμε κατά κάποιο τρόπο μια επιτροπή του Κοινοβουλίου. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί, να ακούμε όλες τις ομάδες και να μην είμαστε μεροληπτικοί. πρέπει να είμαστε ανεξάρτητοι από όλε τι ομάδε, αλλά φυσικά και θα εξαρτώμαστε με την έννοια ότι θα του ακούμε και θα προσπαθούμε να διασφαλίζουμε το συντονισμό μεταξύ του Κοινοβουλίου, αυτή της επιτροπή και του εν λόγω οργανισμού. Σε ό,τι αφορά τώρα την κυρία Λενουάρ. Μιλήσατε για την ανέχεια. Και είναι αλήθεια ότι οι ανισότητες στον τομέα της υγείας εξαρτώνται και από την ανέχεια σε μεγάλο βαθμό. Αν δούμε ποιος είναι ο στόχος και αποστολή του Eurofound, θα δούμε ότι το θεμελιώδες θα πρέπει να είναι να προσφέρουμε υπηρεσίες για την εκπόνηση μελλοντικών πολιτικών, ερευνητικών εργασιών, να διευκολύνουμε τον επιμερισμό και την ανταλλαγή της γνώσης και επίσης να εργαστούμε για να δώσουμε τη δυνατότητα στο Κοινοβούλιο να μπορέσει να νομοθετήσει για την καταπολέμηση των ανισοτήτων. Και όπως είπαμε μπορείτε να ζητήσετε να γίνουν και συγκεκριμένες έρευνες, συγκεκριμένες εργασίες. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό για όλα τα μέλη αυτής της Επιτροπής. Γιατί όπως είπα στην παρέμβασή μου, έχουμε πολλές θεωρίες αλλά μας λείπει η πράξη και από τους οργανισμούς μπορούμε να έχουμε αυτή την πράξη. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε με τον κύριο Μίξιτς. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο να απαντήσω στον κύριο Λένερς καταρχήν. Νομίζω ότι ακριβώς ε, αυτή η τεκτοθεσία ανεξάρτητη πυρογνώμονες που διορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ουσιαστικά ε, λέει πολλά. Θα αναφερθώ συγκεκριμένα εγώ για την όσα. Αυτό εμπλουτίζει τους οργανισμούς. Στον όσα η δομή του Συμβουλίου ουσιαστικά δεν μπορεί να ακολουθήσει τις εξελίξεις της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Όπως σας είπα, υπάρχουν σημαντικές ομάδες πολιτών, μεγάλες ομάδες πολιτών που δεν έχουν άμεση φωνή εκεί στο Συμβούλιο του όσο έχουμε τους εργοδότες, τους εργαζομένους και τις εθνικές κυβερνήσεις. Αλλά έχουμε τόσες πολλές ομάδες, κατηγορίες πολιτών με άμεσο ενδιαφέρον στον τομέα που δεν εκπροσωπούνται. Ακριβώς λοιπόν εσείς έχετε την πιο άμεση σχέση με τους πολίτες, με όλους τους πολίτες. Ακριβώς εσείς και με την παρουσία τη δική μας θα έχετε λέγιν και θα μπορέσετε να εκπροσωπήσετε αυτή την ε, σημαντική ομάδα ανθρώπων. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι με αυτό τον πλούτο, αυτός ο πλουτισμός ουσιαστικά έρχεται με το και εμείς ε, είμαστε εδώ εμπειρογνώμονες και φυσικά τίθεται και το θέμα της διοντολογίας. Η διοντολογία είναι να είσαι ανεξάρτητος. Εγώ προσωπικά πάντοτε θα σας λέω την αλήθεια, ακόμη και αν δεν σας αρέσει. Και για να απαντήσω για το θέμα των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. Είναι τόσο ευρύ το θέμα αυτό. Και αυτό πονάει τόσο πολύ, γιατί οι διαφορές εντός της ευρωπαϊκή Ένωσης μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, ειδικά για το συγκεκριμένο θέμα, είναι τόσο μεγάλες. Και επιπρόσθετα, όταν μιλάμε για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, να δούμε τα τελευταία αποτελέσματα του σενάρ, που είναι μάλλον ένα από τα πιο χρήσιμα προϊόντα του όσα θα δούμε ακριβώς πού έγκυται αυτή η ενισότητα. Ελπίζουμε ότι αυτό θα είναι σημαντικό θέμα στην στη διάταξη του όσα. Για μένα, είναι μέσω είμαι δυνατόν πιο ειλικρινής, βγαίνοντα ε, από αυτό το τυπικό, το επίσημο πλαίσιο, για μένα προσωπικά είναι σημαντικό, πολύ σημαντικό ζήτημα. Και ελπίζω ότι όλοι εσείς εδώ θα το προωθήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ και θα ολοκληρώσουμε το γύρο των ερωτήσεων με τον κύριο Κρέμερ. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Μου έγιναν τρεις ερωτήσεις, αλλά να απαντήσω καταρχάς σχετικά με την υποβολή εκθέσεων. Στην αρχή και όλα στις παρουσίασεις μου, αναφέρθηκα στο ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας είναι κομμάτι της αναγκαίας δομής της Ευρωπαϊκής Ενίας Αγοράς. Είναι η αφετηρία θα έλεγα. Και στις ε, συζητήσεις που είχαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπα ότι εάν κάτι τέτοιο είχε δημιουργηθεί στο τέλος δεκαετίας του 80 ή στις αρχές δεκαετίας του 90, τότε δεν θα υπήρχαν πολλές άλλες ε, δομές που πρόκειψαν στη συνέχεια, διότι θα είχαν ενσωματωθεί στην αρχή αυτή. Έτσι, με τη μορφή που έχει τώρα ως ε, πλατφόρμας που αντιμετωπίζει θέματα παράνομης εργασίας, απόσπασης εργαζομένων κτλ. Με την έννοια αυτή, πρέπει να γίνουν πολλά σε αυτήν την πρώτη περίοδο. Πρέπει να στρώσουμε εμεί το δρόμο για τη συνέχεια. Κύριε έτσι ο διάλογος που είχαμε τον ε, τελευταίο 1,5 χρόνο αφορούσε και, για παράδειγμα, τα αποτελέσματα που έχει να δείξει το τμήμα μας. Νομίζω πως ε, το είπα και αυτό στην ε, παρουσίασή μου, στην αρχή, ότι το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη για περισσότερη ενισχυμένη συνεργασία είτε σε αυτόν τον τομέα, είτε στην ανταλλαγή πληροφοριών ή εμπειριών, είτε μέσω των κοινών επιθεωρήσεων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έπειτα, είναι η πρώτη φορά που λέμε ότι όλοι αυτοί οι τομείς πρέπει να εξεταστούν συντονισμένα, οριζόντια. Ήμασταν πάντα μόνοι μας και γι' αυτό είναι σημαντικό να αλλάξει αυτό. Εάν υπάρξει ένα πρόβλημα ή προκύψει κάποιο ανησυχητικό ζήτημα, τότε πρέπει να δουλέψουμε πιο συντονισμένα για να το επιλύσουμε. Τώρα, υπάρχουν σίγουρα πολλά θέματα σχετικά με την επιβολή, τα οποία έχω εξετάσει όλα αυτά τα χρόνια. Να πω ότι η διεθνική συνεργασία, η συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών αρμόδιων αρχών καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα από επιθεωρήσεις εργασίας αλλά και θέματα ενώσεων, όμορων ενώσεων, οι οποίες μεταφέρουν αρμοδιότητες σε εμά έτσι ώστε να ασχοληθούμε με αυτά τα θέματα συμμόρφωσης. Επίσης, σε ό,τι αφορά την εκτίμηση κινδύνου, υπάρχει επιρογνωμοσύνη και αναφέρθηκε από τον κύριο Ντάνιλσον ο συναγερμός, ο μηχανισμός για συναγερμούς όταν αυτό χρειάζεται. Αν δείτε τις αρχικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα παρατηρήσετε ότι είναι αρκετά περίεργο αυτό που προβλεπόταν, ότι θα υπάρχει δηλαδή αυτό το σύστημα συναγερμού και μετά οι κοινωνικοί εταίροι δεν συμπεριλαμβάνονταν στην πρόταση καν. Κύριε Ντάνιλσον, η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας νομίζω οφείλει να καταρτήσει μια διαδικασία για αυτές τις περιπτώσεις που πρέπει να κυνηγήσει. Εδώ υπάρχει κάποια πείρα σε εθνικό επίπεδο. Και οι αρχές μπορούν λοιπόν να δράσουν. Γιατί δεν μπορείς να, βρει, να εντοπίσει ένα πρόβλημα, μια υπόθεση και μετά να πεις εντάξει, ας το στείλουμε αυτό στην Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας. Πρέπει να δούμε τι συνθήκες επικρατούν. Πρέπει να δούμε τα πορίσματα των ερευνών. και εάν η αντιμετώπιση θα είναι δικαστική ή διοικητική. αν υπάρχουν εμπόδια για να λάβουν κανείς πληροφορίες. Και σίγουρα η περίπτωση θα πρέπει να αφορά παραπάνω από μια χώρα, να είναι διεθνική. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κρέμερ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τις υποψηφιότητές σας, για το χρόνο που διαθέσατε. Τώρα, πώς θα προχωρήσουμε. Θα σας αποχαιρετήσουμε, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα έτσι να προετοιμαστούμε και μετά θα ψηφίσουμε. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να κρατήσετε το πεντάλεπτο διάλειμμα και να μην αργήσετε. Να επιστρέψετε στα μηχανήματα ψηφοφορία σε πέντε λεπτά. Διότι μην ξεχνάτε πως οι διερμηνείς πρέπει να δουλέψουν. Ναι, και εγώ έχω ένα πρόβλημα. Δεν έχω το δικό μου μηχάνημα και δεν μπορώ να ψηφίσω. Πρέπει να το συνδέσουν και ίσως ε, χρειαστούν δύο-τρία λεπτά. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να περιμένουμε. Πρέπει να περιμένουμε και τους ε, υπόλοιπους. Έχουμε ένα πρόγραμμα που πρέπει να τηρήσουμε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αρχίσουμε την ψηφοφορία. Σε πέντε λεπτά λοιπόν. Κυρίε και κύριοι, πέρασαν τα πέντε λεπτά. Πολύ γρήγορα πέρασαν αυτά τα πέντε λεπτά, το ξέρω. Και θα ήθελα να συνεχίσουμε με τις ψηφοφορίες. Οι προσκεκλημένοι μας πρέπει να αποχωρήσουν, διότι η ψηφοφορία είναι μυστική. Λυπάμαι, αλλά πρέπει. Λοιπόν, Σας παρακαλώ να αποχωρήσετε. Wir beginnen mit der Geheimen Wahl. Ξεκινάμε λοιπόν με τη μυστική ψηφοφορία. Ελπίζω να έχουν αποχωρήσει όλοι οι υποψήφοι από την αίθουσα, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να αποχωρήσουν οι υποψήφοι, διότι διαφορετικά δεν μπορούμε να ψηφίσουμε. Δεν βλέπω τους υποψήφιους εδώ. Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και ξεκινούμε με τη μυστική ψηφοφορία για τον κύριο Μπέκερ και την Σεντεφόπ. Άρχεται η ψηφοφορία. ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Ο κύριος Μπέκερ εκλέγεται. Σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με την κυρία Φοντάνη Λόπε για την Eurofound. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Η κυρία Βερόνικα Λόπε Φοντάνια εκλέγεται. Συνεχίζουμε. Ο κύριος Μίξιτς για την EU όσα. Άρχεται η ψηφοφορία. Παρακαλώ ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Πολύ ωραία. Ο κύριος Μίξιτς εκλέγεται στην EU όσα. Τελευταίος υποψήφιος, κύριος Κρέμερς για την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Ο κύριος σε εκλέγεται. You left the room. Φύγατε από την αίθουσα. So, Περνάμε στο σημείο 6. Γενικός προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός μικροφώνου το σχόλιο. Ναι, σας φωνάξαμε μέσα όλους. Οι υποψήφοι αποχώρησαν. Όχι, όχι. Πρέπει να περάσουμε στις ψηφοφορίες, διότι έχουμε και πίεση χρόνου, ξέρετε. Προχωράμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Τροπολογία 5653. Ηλεκτρονικά. Eine elektronische Wahl. Die Wahl ist eröffnet. Άρχεται η ψηφοφορία. Παρακαλώ ψηφίστε. Πέντε χιλιάδες εξακόσια πενήντα τρία. Πέρας. Πέντε χιλιάδες εξακόσια πενήντα τέσσερα. Άρχεται η ψηφοφορία. Με συγχωρείτε κύριε. Τη βάλεστα έφτιαξε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε σε ψηφοφορία με ονομαστική κλίση MP 5655 και 5656. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε. 56-60. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 56-62. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Συνεχίζουμε. 56-63. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 56-67. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 56-68. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται και αυτή. 56-78. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε περασε Πέρας. Εγκρίνατε. 56-93. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνατε. 56-87. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 56-89. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 56-89. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Αυτό ήταν. So, nachher sind die... Περνάμε στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Προσοχή συνεδριάσεις στις 14 και 15 Νοεμβρίου. Λήξη της συνεδρίασης.